Colleagues, uh, take your seats, please. So we begin with the adoption of the agenda. If there are no, if there are no objections, the agenda is adopted. Probably... Καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Αρχίζει η συνεδρίαση. Λοιπόν, η σε διάταξη. Δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Εγκρίνεται. Ωραία. Η διερμηνία. Έχουμε εκτός από γκέλικ, ε, μαλτεζικά, κροατικά, Έχουμε ορισμούς ε, εισηγητών και πρόεδρο όσον αφορά την απόφαση για την Eurojust, όσον αφορά την δικαστική συνεργασία με την Eurojust και τη συνεργασία με τη Δανία. Εγκρίνει η Επιτροπή μας τις συστάσεις των συντονιστών, διαδικασία 205, εγκρίνεται. Δεύτερο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Θεωρήσεις μετά το Brexit. Την 1η Απριλίου οι συντονιστές όρισαν το Σεργέ Στάνιστες από τους ελιστές να είναι εισηγητής για το θέμα αυτό. Το EFTD αμφισβήτησε την απόφαση των συντονιστών να αλλάξει ο εισηγητής και ζήτησε να ψηφιστεί στην Επιτροπή μας η απόφαση αυτή και με ονομαστική ψηφοφορία. Οπότε θα κάνουμε αυτήν την ψηφοφορία τώρα αμέσω. Ονομαστική ψηφοφορία, άρθρο 205, πρέπει 12 ευρωβουλευτές να στηρίξουν το αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία. Οπότε τώρα πρέπει να μας το πούν, να σηκωθείτε παρακαλώ. η διανατάσσεως της χειρός, εντάξει. Λοιπόν, επαναλαμβάνω την ερώτηση. Υπάρχει έτοιμη για ονομαστική ψηφοφορία από το EFTD που πρέπει να στηρίξουν 12 ευρωβουλευτές βάσει του άρθρου 208. Εάν θέλετε να γίνει ονομαστική ψηφοφορία, τότε παρακαλώ είτε σηκωθείτε, είτε διανατάσεως της χειρός, μη συζητάτε, αλλά δείξτε μας αν είσαστε 12 που ζητάτε και στηρίζετε μάλλον αυτό το αίτημα. Λοιπόν, η γραμματεία μου ζητάει να επαναλάβω την ερώτηση. Υπάρχει αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία από το EFTD Λοιπόν, με ακούτε, υπάρχει έτοιμα για ονομαστική ψηφοφορία και απαιτείται να στηριχτεί από 12 μέλη, από 12 ευρωβουλευτέ. Αν θέλετε να γίνει ονομαστική ψηφοφορία μετά από αίτημα του FTD, διανατάσσεω τη χερό ή εφόσον σηκωθείτε, πρέπει να δούμε ότι είσαστε 12 που ζητάτε, που στηρίζετε αυτό το αίτημα. 12 Ωραία, υπάρχουν 12. Οπότε θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε αν συμφωνείτε με τη σύσταση των συντονιστών, δηλαδή την αλλαγή των συντονιστών, ψηφίζετε ναι, συν. Αν είσαστε κατά τη σύσταση των συντονιστών, τότε όχι. Αλλά παρακαλώ, όχι πηγαδάκια, ησυχία. Αν είσαστε κατά τη σύσταση των συντονιστών, να μην αλλάξει δηλαδή η εισηγητή, τότε βάζετε πλην ή μπορείτε να κρατήσετε θέση αποχή Αν είσαστε υπέρ τη σύσταση των συντονιστών για αλλαγή εισηγητή, ψηφίζετε συν. Αν είσαστε κατά τη σύσταση των συντονιστών, ψηφίζετε πλην ή αποχή. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. βλέπω... Μια στιγμή, μια στιγμή. Θα βοηθούσε αν με ακούγατε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Γιατί έχουμε τέσσερις παραπάνω από το ΕΛΚ που ψηφίζουν. Τέσσερις επιπλέον από τους σοσιαλιστές. Οπότε παρακαλώ Βγάλτε τις κάρτες από το μηχάνημα όσοι είσαστε επιπλέον. Από τους σοσιαλιστές ένας παραπάνω είναι. Περιμένω. Οι σοσιαλιστές έχουν έναν παραπάνω. Για λύστε το αυτό. Συν τρεις έχουν τώρα οι σοσιαλιστές. Χειροτερεύει το πράγμα. Συν τέσσερις τώρα. Καλά όλη μέρα μα θέλετε θα καθίσουμε εδώ πέρα. Συν ένας σοσιαλιστές πάντα. Μην πειράζετε τίποτα. Είμαστε εντάξει τώρα, πέρα τη ψηφοφορία. 29 υπέρ, 16 κατά και 3 αποχές. Περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία, που είναι το σημείο 3, που είναι η ψηφοφορία για τη συμφωνία. Πριν ψηφίσουμε όμως, ο εισηγητής θέλει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ναι, βεβαίω και πρέπει να πάρω το λόγο, γιατί δεν είναι μια συνηθισμένη κατάσταση αυτή για την Επιτροπή μας. Και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι με όρισαν οι συντονιστές προχτές στις 4 το απόγευμα. Είμαι και αντιπρόεδρος στην Επιτροπή μας. Και πρέπει να σας πω ότι έχοντας κάνει ένα γύρο τριμερούς διαλόγου με την Επιτροπή και το Συμβούλιο, το θέμα δεν είναι ο εισηγητής δεν υπήρξε βούληση από πλευράς του Συμβουλίου να φτάσουμε σε κάποιο συμβιβασμό. Όταν ανέλαβα την αποστολή αυτή, καλή την πίστη, προσπάθησα να διατυπώσω ένα τέταρτο συμβιβασμό εκ μέρου της Επιτροπή μα. Διότι πάντοτε ήμασταν επικοδομητικοί και πάντα ήμασταν υπέρ του πνεύματος συνεργασίας και συμβιβασμού που διέπει την Ευρώπη. Είχαμε και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του 2017 που και ευχαριστώ και τη γραμματεία της Επιτροπής μας που με βοήθησε να καταλήξω σε αυτό το σεβασμό. Προσπάθησα λοιπόν να λάβω υπόψη μου όλες τις απόψεις για το ευαίσθητο θέμα του Γιβραλτάρ. Ευχαριστώ επίσης τους σκιώδες εισηγητές για τη στήριξή τους και την κατανόησή τους, γιατί έπρεπε να βρεθούμε πριν από αυτό τον τελευταίο έκτο τριμερή διάλογο και να καταλήξουμε σε ένα κοινό τόπο για να πάμε στη συνέχεια στο Συμβούλιο. Είναι σημαντικό να δείξουμε ότι η Επιτροπή μας θέλει μία λύση. Μετά όμως από αυτή τη συνάντηση μπορώ να σας πω ότι ο πρόεδρος μας, ο κύριος Κλοντ Μωράης, είχε εξαιρετικές διαπραγματεύσεις στους πέντε πρώτους γύρους, έκανε ό,τι μπορούσε, ε, πρότεινε τρεις διαφορετικές συμβαστικέ προτάσεις, η δικιά μου ήταν η τέταρτη, αλλά δεν υπήρξε βούληση καθόλου από πλευρά του Συμβουλίου, ό,τι και αν κάναμε. Αυτά προς ενημέρωσή σας. Όμως υπάρχουν και δύο ακόμα πράγματα. Το ένα είναι η ίδια η ζωή. Ένα πράγμα που δεν μπορούμε να αρνηθούμε είναι ότι φτάνει ολοταχώς η 12η Απριλίου και παίζεται εκεί η τύχη εκατομμυρίων ε, Βρετανών και πολύ περισσότερων εκατομμυρίων ε, Ευρωπαίων που θα ταξιδεύουν ή όχι με θεώρηση. Το δεύτερο θέμα είναι η υπευθυνότητα, γιατί η στρατηγική του Συμβουλίου στις διαπραγματεύσεις αυτές ήταν λιγάκι μια στρατηγική που ήθελε να πάνε τα πράγματα στα άκρα και μετά να λυγίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα προτείνω να στηρίξετε την έκθεση γιατί η δικιά μας ευθύνη είναι πολύ μεγαλύτερη από το απλώς να τσακωνόμαστε μεταξύ μας και ένας να κατηγορεί τον άλλον και να λέμε να αυτοί φταίνε. Οι Βρετανοί και οι Ευρωπαίοι ε, πρέπει να μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς τόρους. Εμείς δεν μπορούμε να αφήσουμε την πρόταση αυτή χωρίς να τη στηρίξουμε. Ε, δεν περίμενα ότι θα πρέπει να λάβουμε το λόγο γιατί και το Συμβούλιο βρίσκεται σε μία ε, μεταβατική κατάσταση ε, και γι' αυτό κύριε Σάνιτσεφ ανέκεψε αυτό το ζήτημα. Δυστυχώς όμως θα πρέπει να δούμε όλα τα σημεία, τα διαδικαστικά που εθίγησαν από την ομιλία σας. Άρα ή θα λάβουμε υπόψη όλες τις ομιλίες, αλλά επειδή έκανε μία ομιλία ο εισηγητής, έχουμε και άλλους ομιλητές, τους οποίους θα πρέπει να ακούσουμε εφόσον ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία. Ε, ε, δεν, έχει ε, λόγο, δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή να με επιπλήτετε, γιατί αλλιώς θα μιλήσω κι εγώ. Ναι, συγγνώμη, προεδρεύω. Κανένας δεν προεδρεύει από άλλες επιτροπές. Υπομονή και ησυχία. Έχουμε πολλά σημεία από τα μέλη. Μπορείτε να γνέφετε αρνητικά, αλλά η ουσία είναι ότι ανακύπτουν ζητήματα από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Εάν θέλουν να λάβουν το λόγο, μπορούν. Κυρία Ιντβέλτ, διαδικαστικό. Εντάχει, καταρχήν να σας ευχαριστήσω γιατί το επιτρέπετε. Θεωρώ ότι θα πρέπει να εκφράσω τις απόψεις μου πριν ψηφίσω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον νέο εισηγητή για τα λόγια του. Ήταν ακριβέστατος. Εγώ θα υπερψηφίσω την έκθεση για τους λόγους που προανέφερε ο εισηγητής αλλά ο τρόπος από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο με αφήνει με μια άσχημη, ε, ε, με άσχημη γεύση. Ευχαριστώ πολύ. Έχω ένα διαδικαστικό, λέει ο κύριος ε, Ζούλιστρα ο Ολλανδός Υπουργό, ο οποίος ήταν ε, υπεύθυνος για τις διαπραγματεύσεις, ερωτήθη χτες γιατί υποστήριξαν οι Ολλανδοί το θέμα σε έξι στο Συμβουλίο. Είπε ότι όχι, σιωπήσαμε, γνωρίζουμε ότι το ε, κείμενο προσαρμόστηκε και όταν ε, ερωτήθη ποιο είναι το προσαρμοσμένο κείμενο διάβασε ακριβώς το ίδιο και είπε ότι αυτή είναι η τελευταία νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η οποία δεν είναι. Άρα ήταν κακώς πληροφορημένος ο Ολλανδός υπουργό και νομίζω ότι το Συμβούλιο δεν ε, διαπραγματεύτηκε καλή την πίστη. Υπήρξε κακή εκπροσώπηση στις έξι συναντήσεις και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη κατά την ψηφοφορία, τουλάχιστον εγώ θα το λάβω. Η κυρία Ρίτ, δυνάμει του 2-6, όπως και ο κύριος Κάρβερ, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, η θέση να αποσύρουμε έναν ε, ευρωβουλευτή από την έκθεση αυτή σε σχέση με το Γιβραλτάρ και τη θέση του, Ε, το ότι ζητήθηκε να αποσυρθεί Βρετανός Ευρωβουλευτής και να μπει κάποιος άλλος λόγω του θέματος του Γιβραλτάρ είναι κάτι το απαράδεκτο. Δυνάμει της ε, ε, χάρτας των Ηνωμένων Εθνών είναι ένα μια αυτόνομη επικράτεια το Γιβραλτάρ και δεν έχει νόημα, είναι απαράδεκτο να αμφισβητήσετε την κυριαρχία του Γιβραλτάρ. 52 χρόνια πριν, το 99% των κατοίκων του Γιβραλτάρ ζήτησαν να παραμείνουν υπό την αιγίδα του Ηνωμένου Βασιλείου και παρόμοια αυτό επικράτησε το 2002 ως μία ευρωβουλευτή η οποία βρέθηκε στην επέτειο, στην πετικοστή επέτειο, θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο αυτή η θέση. Πρέπει να σας διακόψω, κυρία Ρίντ, λέει ο πρόεδρος. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη η απόφαση των συντονιστών. Κάρβερ, εντάχει. Ο η συγητή μίλησε για γεγονότα τη ζωή. Μην ξεχνάμε ότι γίνονται εκλογέ στην Ισπανία σύντομα και μιλάμε για την εσωτερική πολιτική της Ισπανίας εδώ. Νομίζω ότι είναι ε, απαράδεκτο να λαμβάνουμε υπόψη θέματα μικροπολιτικής για να λαμβάνουμε αποφάσεις. Κάποιος άλλος όχι, άρα ψηφίζουμε. Γίνονται συζητήσεις βλέπω, θα ήθελα όμως να μην γίνονται, γιατί ο κύριος ε, Τζέζα και άλλοι δεν είναι παρόντες. Ε, εγώ δεν θα ήθελα να θίξω παρεμφερή ζητήματα. Δεν θα ήθελα να μιλήσω για την ακαιρεότητα του Κοινοβουλίου, τη συμπεριφορά του Συμβουλίου έναντι του Κοινοβουλίου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ας ε, είμαστε αξιοπρεπείς, ας περάσουμε στην ψηφοφορία η οποία και άρχεται. Ε, τρεις υπεράριθμοι από το ΕΛΚ, παρακαλώ να βγάλετε τις ε, κάρτες σας. ΕΛΚ συν 2, σοσιαλιστές συν 2, σοσιαλιστές συν 1 υπεράριθμος. Πέρας. 34, ε, 8 κατά και 3 αποχές. Και 8 αποχές, όχι 3 αποχές, με συγχωρείτε, 38, 8, 3. Λήξη της ψηφοφορίας.